ξεκινήσουμε χωρίς να χάνουμε πολύ χρόνο. Όσο κάθεστε θα διεκπαιρώσω εγώ τα τυπικά. Πρώτα απ' όλα έγκριση της μέρσιας διάταξης. Δέχεστε την μέρσια διάταξη, δεν βλέπω να ζητά κάποιο το λόγο, άρα η μέρσια διάταξη γίνεται δεκτή. Σημείο 2 έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 21ης Ιανουαρίου και 10ης Μαΐου. Σίγουρα. Σίγουρα. μάλιστα. Περνάμε στο επόμενο. Απλά είχαμε μείνει λίγο πίσω στα πρακτικά, γιατί λέω και εγώ από το Γενάρη έχουμε να πρακτικά. Λοιπόν, ανακοινώσεις. Πρώτα απ' όλα, εάν δεν υπάρχουν αρκετά έδρανα, υπάρχει και μία αίθουσα στην οποία μπορείτε να ακούσετε Γιάν 2Q2. Μπορείτε να ακούσετε τη συνεδρίαση από εκεί. Δεύτερη ανακοίνωση. Σύμφωνα με τον κανόνα 73, μάλλον 70 σημείο 3 ε, του κανονισμού, πρέπει να σας πω ότι διαπραγματεύσεις ε, για την πρόταση AMFMD ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και οδήγησαν λοιπόν σε μια συμβιβαστική λύση με το Συμβουλίο. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκοζέ, στον εισηγητή, μετά την ανταλλαγή απόψεων τον κύριο Γιούγκερ, για να μας ενημερώσει. Αυτό θα γίνει γύρω στις 4 και 30 σήμερα. Εάν λοιπόν θέλει κάποιος από εσάς να εκφράσει τις απόψεις του και να ακούσει τα σχετικά, θα πρέπει να παραμείνει. Επίσης, μπορώ να σας πω ότι υπάρχει μια έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου, στο Στρασβούργο δηλαδή έχει προγραμματιστεί ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Μπαρνιέ στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου που είναι σε εξέλιξη και ελπίζουμε να έχουμε ανταλλαγή απόψεων και με τον Επίτροπο Ρέν για να συζητήσουμε το έργο σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου. Τέλος, θα ψηφίσουμε την έκθεση Γκοζές για, τις, ε, για τους οίκους αξιολόγησης. Ε, αναβλήθηκε για αύριο και 22 Νοεμβρίου στην έκτακτη συνεδρίαση θα γίνει αυτό. Σημείο 4. Να καλωσορίσω και πάλι με πολύ μεγάλη χαρά τον κύριο Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ, πρόεδρο του Eurogroup, ο οποίος ως συνήθως θα μας κάνει έναν απολογισμό της κατάστασης εντός ευρωομάδας και θα επακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων με τους βουλευτές Μέρο το οποίο και ο ίδιος ο κύριος Γιούνκερ έχει πει ότι θεωρεί και το πιο ενδιαφέρον στην όλη διαδικασία. Κύριε Γιούνκερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, αγαπητοί φίλοι, είναι πάντα με μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι ενώπιον σας μετά από μια αρκετά μεγάλη απουσία για να σας ε, αναφέρω ε, και να αναφερθώ σε διάφορα θέματα που μας απασχολούν όλους μας και απαιτούν ε, ιδιαίτερη προσοχή. Ήδη ευθύς εξ αρχής θα πρέπει να σας πω ότι προφανώς μετά από αυτή την άνευ οικονομική κρίση που διανύουμε ε, είμαστε πάντοτε αντιμέτωποι με μια κατάσταση όλο και πιο δύσκολη σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στο ευρωπαϊκό επίπεδο και διαβάζω παντού ότι ναι, βγαίνουμε από τα επικίνδυνα νερά, ναι, ότι βλέπουμε το φως στην άκρη του τούνελ. παρόλα αυτά όμως έχουμε ένα αρκετά μικρό ε, ποσοστό ε, μεγέθησης. Ε, στα πλαίσια της ζώνης του ενιαίου νομίσματος. Ε, το ποσοστό αυτό είναι σαφώς κάτω από το επίπεδο που θα έπρεπε να βρίσκεται αν είχαμε ε, βρει τους ρυθμούς ανάπτυξης που είχαμε πριν από την έναρξη της κρίσης αυτής. Θα πρέπει όλα λοιπόν να γίνουν ούτω ώστε μέσα από τις ε, απαραίτητες διαρθρωτικές ε, μεταρρυθμίσεις να ξαναβρούμε το ρυθμό ανάπτυξης ε, που χρειάζεται η ζώνη. Είναι γεγονός ότι συμφωνήσαμε και στο επίπεδο των G20 και στο επίπεδο της Ευρωζώνης για τον τρόπο εξόδου από την κρίση που θα αρχίσει αργότερα ε, το 2011 ε, με τα φορολογικά ε, κίνητρα. Υπάρχουν πάντως κάποιοι καθολικοί στόχοι που πρέπει να επιτύχουμε. Η εξυγίαση πρώτα απ' όλα είναι ο στόχος μας, η εξηγίαση των δημόσιων οικονομικών και του δημόσιου χρέους. Αλλά χρειάζεται κάποια προσοχή σχετικά με τα μέτρα που θα χρησιμοποιήσουμε, ούτε ώστε να μην ε, υπερβάλλουμε ε, σε αυτά που κάνουμε και εφαρμόσουμε έτσι πολιτικές που θα μπορούσαν να είναι εις βάρος της ανάπτυξης. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ιδιαίτερα προβλήματα σε ορισμένες χώρες. Θα σας μιλήσω για την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα. Εγώ πάντοτε θαυμάζω τη σοβαρότητα και την ποιότητα των αντεδράσεων των Ιρλανδικών αρχών ε, που όπως ξέρετε στις 4 Νοεμβρίου ανακοίνωσαν μια συμπληρωματική προσπάθεια οικονομικής εξυγίανσης που αφορά 6 δισεκατομμύρια ευρώ το διπλάσιο δηλαδή του ποσού που είχαν ανακοινώσει οι Ιρλανδοί φίλοι μας πριν από τρεις μήνες. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια και θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής στις κυριότερες ε, ε, Ιρλανδικές πολιτικές δυνάμεις που συμφώνησαν στα κύρια σημεία ε, των όσων θα πρέπει να γίνουν και συμφώνησαν πάνω σε κοινά μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν είμαι πεπισμένος ότι οι Ιρλανδικές αρχές θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν στην πράξη αυτό το πολιετές ε, πρόγραμμα εξυγένσης που είναι τετραετές, ούτως ώστε η διόρθωση του ελλείμματος το 2014 να ε, ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας. Και είμαι πεπισμένος ότι οι συνδυασμένες προσπάθειες όλων των ε, εμπλεκομένων στην Ιρλανδία θα ε, μπορέσουν να βάλουν τη χώρα αυτή που δοκιμάζεται τόσο σκληρά ε, στο δρόμο της ε, βιώσιμης της αηφόρου ανάπτυξης. Ίδιες παρατηρήσεις για την Πορτογαλία, όπου και εδώ πάλι θα πρέπει να τιμήσω και την κυβέρνηση και τα ε, μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης που συμφώνησαν όσον αφορά το δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσουν. Ξέρετε, όπως και εγώ, ότι ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε κατά την πρώτη ανάγνωση ε, στις 3 Νοεμβρίου στο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, στο Πορτογαλικό Κοινοβούλιο. Η δεύτερη ανάγνωση θα γίνει γύρω στις 26 Νοεμβρίου και πιστεύω ότι και εδώ έχουμε βάσιμους λόγους να ε, είμαστε πεπισμένοι ότι οι πορτογαλικές αρχές θα επιτύχουν να περάσει ο προϋπολογισμός για το 2011 από το Κοινοβούλιο και δεν θα αργήσει η Πορτογαλία να ξεκινήσει τις ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται τόσο ώστε ε, το αναπτυξιακό δυναμικό της ε, Πορτογαλίας να διορθωθεί προς τα πάνω. Δεύτερη ζώνη που προκαλεί ανησυχίες είναι η Ελλάδα. Και εδώ πάλι ξέρετε ότι θα ανακοινωθούν αριθμητικά στοιχεία που θα αφορούν τον προϋπολογισμό και το χρέος, που θα καθορίσουν στη συνέχεια αυτά που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο καιρό. Και εδώ όμως δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανησυχία. Πιστεύουμε ότι οι ελληνικές αρχές θα είναι σε θέση να σεβαστούν ε, με μια προοπτική του 2014 ε, τους, τις δημοσιονομικές διορθώσεις που έχουν ε, αποφασιστεί. Και πιστεύω επίσης ότι οι ελληνικές αρχές θα είναι σε θέση να τηρήσουν και να επιτύχουν και τους στόχους που έχουν τεθεί για το 2011. Γενικότερα όσον αφορά το μηχανισμό στήριξης για την Ελλάδα, δεν θέλω να σας κάνω μια ε, αναλυτική παρουσίαση, γιατί τα ξέρουμε όλα αυτά απ' έξω. Πιστεύουμε ότι το αυστηρό ε, πρόγραμμα το οποίο αποφάσισε η ελληνική κυβέρνηση είναι αξιόπιστο και παραμένει αξιόπιστο και θα μεταφραστεί σε συγκεκριμένα γεγονότα. Ξέρετε ότι θα πραγματοποιείτε κάθε τρεις μήνες ε, διάμεση ε, επανεξέταση και έκθεση. Ε, έγινε αυτό πριν από την απελευθέρωση της πρώτης δόσης που αφορούσε 18 δισεκατομμύρια τον Μάιο και μία δεύτερη που αφορούσε 6,5 δισεκατομμύρια τον Σεπτέμβριο. Παρ' όλα αυτά, ε, ισχύει και παραμένει το γεγονός ότι η ανάπτυξη στην Ελλάδα έχει υποχωρήσει όπως και το 2010 και άρα η, ε, θα πρέπει να δούμε τι θα δώσουν οι, μεταρρυθμι... οι... Ε, οι δομικές μεταρρυθμίσεις και να δούμε αν θα χρειαστεί ενδεχομένως να, λάβει η ελληνική κυβέρνηση και πρόσθετα μέτρα, ούτως ώστε να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι, οι δημοσιονομικοί στόχοι. Ε, δεν έχω πολλά να προσθέσω. Σχετικά με τις ε, ανησυχίες σχετικά με τον, ε, το EFSF, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό ε, ε, ε δημοσιονομικής στήριξης, ο οποίος αποφασίστηκε στις 7 Μαΐου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στη συνεδρία του ΕΚΟΦΗΝ στις 9 Μαΐου. Αυτά είναι λειτουργικά ήδη από τον Ιούλιο. Δεν ξέρω, κυρία Πρόεδρε, αν σας δόθηκε η ευκαιρία να έρθετε σε επαφή με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, του, ε, τον κύριο Κλάους Ρίκλινγκ, μιας εταιρείας που η έδρα της είναι στο Λουξεμβούργο. Αν δεν σας δόθηκε μέχρι τώρα η ευκαιρία, θα σας πρότεινα να τον ε, προσκαλέσετε τον κύριο Ρίγκλινγκ, ώστε να σας εξηγήσει ε, με κάθε λεπτομέρεια το μηχανισμό αυτό και τον τρόπο με τον οποίο θα δοθεί συνέχεια στις αποφάσεις ε, της ε, Ευρωζώνης. Ο κύριος Ρίγκλινγκ ε, θα σας δώσει όλες αυτές τις πληροφορίες και αν μου επιτρέπετε θα σας πρότεινα να οργανώσετε μία ειδική ακρόαση για να ακούσετε τον κύριο Κλάους Ρίγκλινγκ. Αλλά είμαι και εγώ βέβαια στη διάθεσή σας για να σας δώσω και εγώ ό,τι απαντήσεις ενδεχομένως θέλετε. Ήδη εδώ και αρκετούς μήνες ανακοίνωσα ότι θα ξεκινήσουμε μια ειδική ε, εργασία μέσα στην Ευρωζώνη, δηλαδή ότι θα παρακολουθήσουμε πολύ πιο προσεκτικά τις μακροοικονομικές ανισορροπίες που υπάρχουν στα διάφορα κράτη-μέλη της ζώνης. Ε, πιστεύουμε πραγματικά ότι δεν ε, δώσαμε αρκετή προσοχή στις διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, διαφορές που παραμένουν, που είναι μεγάλες, είναι μεγάλες διαφοροποιήσεις και άρα θεωρούμε ότι είναι καθήκον μας να μετατρέψουμε σιγά σιγά την ε, ε, νομισματική ζώνη του ευρώ σε μια ζώνη που να λειτουργεί ε, με καλύτερο τρόπο, με τον στο δυνατό τρόπο. Άρα θα πρέπει να κάνουμε ό,τι δυνατόν για να ε, απαλείψουμε τις μακροοικονομικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών. Ξεκινήσαμε μια άσκηση peer review για κάθε χώρα δηλαδή της Ευρωζώνης εξετάσουμε πολύ πιο προσεκτικά τους δείκτες, τις διάφορες υποζώνες, διάφορες μέρου ζώνες της Ευρωζώνης. Εξετάσαμε Ισπανία, Φιλανδία, Πορτογαλία και Λουξεμβούργο την τελευταία περίοδο. Κατά την επόμενη περίοδο θα εξετάσουμε πιο λεπτομερώς τη κατάσταση στη Γερμανία και στην Ιταλία. Και τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε δεν έχουν τίποτα το ε, περίεργο, γιατί σε κάθε μία από τις χώρες που εξετάσαμε και που θα εξετάσουμε, διαπιστώνουμε την ανάγκη περιορισμού του διαρθρωτικού ε, ελλείμματος που παρουσιάζουν οι εθνικοί προϋπολογισμοί, οι κρατικοί προϋπολογισμοί και ε, κάνοντας κάτι τέτοιο θα εξασφαλίσουμε μια αυξημένη αξιοπιστία. Διαπιστώνουμε ε, επίσης από την εξέταση των διαφόρων κρατών μελών ότι ε, ένας ιδιαίτερος κίνδυνος προκύπτει από το υψηλό επίπεδο του δημόσιου χρέους. Ε, υπάρχει μεγάλη χρέωση και των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και αυτό είναι απαραίτητο να περιοριστεί για να αποευθούν μελλοντικές φούσκες. Κατά τα άλλα, ε, θα εξετάσουμε περισσότερο την κατάσταση στην αγορά εργασίας που εξακολουθεί να παραμένει άσχημη και κάποιες ε, ε, ε, αρνητικές πτυχές της διαμόρφωσης των μισθών στην ζώνη του ευρώ. Δυσκολίες λοιπόν στην αγορά εργασίας, ακαμψία στην αγορά εργασίας που είναι πολύ μεγάλη και μεταφέρεται από τη μια χώρα στην άλλη. Ακαμψία λέω, αναλαστικότητα της αγοράς εργασίας που δεν διορθώνεται γιατί ε, συνεχίζουν ε, πολλοί να διαμαρτύρονται για τις ε, των ε, εργοδοτών. Το γεγονός λοιπόν ότι λέμε ότι θα πρέπει να ε, διορθωθεί το θέμα της ελαστικότητας, της ανελαστικότητας της αγοράς εργασίας δεν σημαίνει ότι ε, ζητάμε από τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν ή να αρχίσουν να εφαρμόζουν όπου δεν υπάρχει αυτή την αχαλήνοτη, ε, την ε, αυθαίρετη θα λέγαμε ελαστικότητα. Θέλουμε καλές πολιτικές και όχι οποιαδήποτε πολιτική που να κινείται πίσω από τον ε, τίτλο της ελαστικότητας αγοράς εργασίας και να καταλήγει σε υπερβολές. Πέραν αυτού δεν έχω πολλά πράγματα να σας πω. Να σας θυμίσω απλώς ότι έχουμε ένα κοινό διάβημα που ε, ξεκινήσαμε ε, στην Ευρωομάδα. Ε, συνεχίζουμε δηλαδή να λέμε ότι δεν θέλουμε αυτή την ε, εξαιρετική μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών. θεωρούμε ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να εξασφαλίσουμε τα απαραίτητα χρηματοοικονομικά δεδομένα και ότι δεν θα πρέπει να οδηγηθούμε σε εθνικές συμπεριφορές που να βασίζονται σε εγωιστικές αντιδράσεις και δεν θα πρέπει ε, οι διεθνείς αγορές να ε, ε, χάσουν την, το ρόλο τους. Η G7 φυσικά δεν θα πρέπει να εξαφανιστούν ε, και πρέπει να σας πω ότι ένας Λουξεμβούργιος, για να πω κάτι το αυτοβιογραφικό, για πρώτη φορά κατάφερε να διεισδύσει στους G7, στους Υπουργούς ε, Οικονομικών και μόλις οι Αμερικάνοι έμαθαν ότι πήγαινα εκεί, άλλαξαν τον ε, χώρο της συζήτησης και η πραγματική συζήτηση γίνεται πια στο επίπεδο των G20. Θα δούμε τι θα αποδώσει αυτή η αλλαγή, αλλά έχω πραγματικά ε, την ελπίδα ότι η G20 θα αποδειχθεί ότι θα είναι η παγκόσμια δομή όπου θα μπορέσει πραγματικά να συζητηθεί το θέμα των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ε, είχα παραστεί πολλές φορές στις συνεδριάσεις των G7 και πρέπει να σας πω ότι όταν τα θέματα συζητούνται στο επίπεδο τον G20 ο μεγάλος κίνδυνος είναι να μην κάνουν τόσο έντονη ανταλλαγή απόψεων οι 20 όπως γινόταν στο επίπεδο των G7. Ε, και μετά τις συνεδριάσεις των G20, ε, στις εφημερίδες θα, μάθουμε, ε, θα μάθουν αυτοί που δεν ζητήθηκε η γνώμη τους όπως των άλλων. Οι Financial Times λένε πάντα τι συμβαίνει σε αυτές τις συνεδριάσεις και ενημερώνουν αυτούς που δεν παρευρέθηκαν. Εν πάση περιπτώσει, είναι μεγάλη ευκαιρία αυτή για να διευρυνθεί ο κύκλος αυτών που συμμετέχουν στη συζήτηση. Γιατί οι αναδυόμενες χώρες, οι ασιατικές χώρες, η Βραζιλία και άλλες ε, θα πρέπει να έχουν ε, λόγο, δικαίωμα λόγου ε, για τα θέματα αυτά. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι η Ευρωομάδα δεν εκπροσωπείται στη δομή των G20 κάποια μέρα όταν θα γράψω τα απομνημονεύματά μου θα σας εξηγήσω και τους επιφανειακούς και τους βαθύτερους λόγους για τους οποίους η Ευρωομάδα ε, ε, δεν συμμετέχει στους ε, G20. Δεν είναι όμως φυσιολογικό η Ευρωομάδα να εκπροσωπείται μόνο από τον Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ εμείς επί <clears throat> ώρες ατέλειωτες ακούμε όλες αυτές τις διαλέξεις για την ενίσχυση του ρόλου μας κλπ. Δεν είναι θέμα λοιπόν της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά της Ευρωομάδας. Όταν συζητάμε την οικονομική πολιτική, ε, η Ευρωομάδα εκπροσωπείται από τον διευθύντη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ενώ επί σειρά ετών εξηγούμε ότι το λάθος της οικοδόμησης της Νομισματικής Ένωσης είναι ότι ευνοήσαμε την νομισματική πτυχή ε, σε σχέση με την πολιτική, την νομισματική διάσταση σε σχέση με την πολιτική διάσταση. <clears throat> Αλλά θα πρέπει να ρωτήσετε αυτούς που φαντάστηκαν αυτή την χορογραφία των G20, αυτή την ε, δομή τέλο πάντων, χωρίς ε, εκπροσώπηση της ευρωομάδας. Και ακόμα πιο γελίο θεωρώ ότι κανένας ε, στην Ευρώπη δεν έχει την πιθανότητα να επιτύχει αλλαγή ε, στους G20 ώστε η Ευρωμάδα να βρει εκεί τη θέση της. Σε επίπεδο δομών της Ευρωμάδας και του ΕΚΟΦΗΝ και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ε, έχουμε τρόπο να ασχοληθούμε με τους G20. Το κάναμε αυτό και στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και πρέπει να σας πω ότι είναι μια συζήτηση αρκετά σύντομη. Πράγμα το οποίο με κάνει να ε, υποθέσω ότι συμφωνούμε ε, σε όλα τα σημεία που δεν αναφέρθηκαν. Πιστεύουμε αυτή τη στιγμή ότι το δολάριο σε σχέση με το ευρώ δεν βρίσκεται στο επίπεδο στο οποίο θα έπρεπε να βρίσκεται. Οι πρόσφατες αποφάσεις της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας δεν μου φαίνεται ότι ανταποκρίνονται σε όλες τις προσδοκίες που τρέφαμε εμείς ε, από πλευράς Ευρωπαϊκής Νομισματικής Πολιτικής. Βλέπουμε περισσότερους κινδύνους και ε, δυσκολίες ε, σε παγκόσμιο επίπεδο μετά από τις αποφάσεις αυτές που έλαβε η ΦΕΔ που επιστημονικά ίσως είναι ε, βάσιμες, αλλά θα δούμε κατά τις προσεχείς εβδομάδες και μήνες τι ακριβώς θα δώσουν. Αλλά ξεκινάμε από την αρχή ότι ε, οι Ευρωπαίοι ε, που θα βρεθούν γύρω από το τραπέζι των G20 δεν θα παραλείψουν να θέσουν ερωτήματα στους Αμερικάνους φίλους μας σχετικά με τις πρόσφατες νομισματικές τους αποφάσεις που δεν είναι καθόλου ευθυγραμμισμένες ε, με αυτά που αποφασίστηκαν στις ε, παρασκευαστικές εργασίες των G7 και των G20. Τώρα για την διακυβέρνηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν θα πω πολλά πράγματα. Θα πω ε, μόνο ότι συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι υπάρχουν πολλοί λαγοί γύρω από το τραπέζι των, ε, ε, του Δούνου του. Από τους 26-7 είναι οι Ευρωπαίοι. Υπάρχει μια ευρώ... Ε, ε, υπεροψία ε, πέραν των επιτρεπτών ε, επιπέδων και γι' αυτό πρέπει να γίνει κάποια διόρθωση από πλευράς Ευρώπης. Εγώ πάντοτε θεωρούσα ότι η ζώνη του ευρώ θα πρέπει να εκπροσωπείται στα όργανα των διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών, αλλά μόνο με μία έδρα. Αυτός ήταν ο στόχος μας. Ο κύριος εταίρος σήμερα είναι ο Αμερικάνος βέβαια στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αλλά και οι Ευρωπαίοι που εξελίσσονται γύρω από την Ευρωζώνη δεν βλέπουν ποιος είναι ο λόγος ή το συμφέρον να συγκεντρωθούν γύρω από τα ε, ευρωπαϊκά συμφέροντα. Ε, λυπάμαι που είναι έτσι τα πράγματα, αλλά αυτό δείχνει η ιστορία. Ήδη το άρθρο 138 της συνθήκης δείχνει ε, ότι η Κομισιόν θα πρέπει να απευθύνει στο Συμβούλιο μία πρόταση που θα έχει σαν σκοπό να βελτιώσει την ε, εκπροσώπηση στο εξωτερικό της ε, ζώνης του ευρώ. Η ιστορία κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς χάνουμε χρόνο, οι άλλοι αποφελούνται από αυτό, ε, χαίρονται να βλέπουν τους Ευρωπαίους να κατασπαταλούν την δυνατότητα επιρροής που έχουν εδώ και εκεί, αντί να επικεντρώνουν τις δυνάμεις τους την ευρωπαϊκή επιρροή. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν υπερβολικά πολλοί Ευρωπαίοι στο τραπέζι του Δουνουτού και όχι αρκετή Ευρώπη. Και, πρέπει, πιστεύω ότι, και πιστεύω ότι πρέπει οι Ευρωπαίοι να υποφεληθούμε από τη μεταρρύθμιση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ώστε να έχουμε μεγαλύτερη επιρροή εκεί μέσα. Σε ό,τι αφορά τώρα την ομάδα εργασία του Χέρμαν και για τα πρόσφατα αποτέλεσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μπορώ να σας ενημερώσω εν συντομία. Συμφωνήσαμε για τα στοιχεία της μεταρρύθμισης ε, του Συμφώνου Σταθερότητας Και φυσικά όχι μόνο γιατί μας υποχρώνει συνθήκη. Η μεταρρύθμιση αυτή και τα διαφορετικά της στοιχεία γίνονται σε στενή συνεννόηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βέβαια, δεν είναι η σωστή λέξη αυτή που χρησιμοποιώ και δεν θα έπρεπε να μιλώ για συνεννόηση, αλλά για συναπόφαση. Θεωρώ προφανές ότι όταν μιλάμε για την ε, σταθεροποίηση των οικονομικών, όταν θέλουμε οι δημοσιονομικές προοπτικές της Ευρωζώνης να δουν καλύτερες ημέρες και καλύτερους ιονούς. Θεωρώ δεδομένο τα δύο σκέλη της, ε, του προπολογισμού, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο, θα πρέπει να βαδίζουν προς την ίδια κατεύθυνση. Θα πρέπει να το γνωρίζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όταν συναντηθήκαμε πρόσφατα είχα υπενθυμίσει ότι το Κοινοβούλιο όχι μόνο έχει λόγο, να πει, αλλά πρέπει και να συναποφασίζει. Πάνω σε αυτό λοιπόν θέλω να σας πω ότι μιλώντας εγώ προσωπικά, έχω να πω τρία πράγματα. Δεν έχω εντολή ε, από την Ευρωμαδία να τα πω αυτά. Λοιπόν, πρώτον, θεωρώ ότι οι αποφάσεις για τις κυρώσεις πρέπει να είναι ακόμη πιο αυτόματες σε σχέση με αυτό που ε, αποφασίστηκε στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι η αρχική πρόταση της Κομισιόν δεν ανταποκρινόταν, δεν αντιμετώπιζε όλα τα προβλήματα που ετίθεντο Δηλαδή, δεν μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι αποφασίζει μόνο η Κομισιόν και εκτελούν τα κράτη-μέλη. Φυσικά πρέπει να υπάρχει ένα στοιχείο πολιτικής κρίσης. Πολιτική κρίση λοιπόν που θα εκφράζεται από το Συμβούλιο. Δεν επαρκεί επίσης να προβλέπουμε την αντίστροφη ειδική πλειοψηφία για την επιβολή κυρώσεων. Θα έπρεπε να αποφασίζουμε πάντοτε με την ειδική πλειοψηφία, την ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας που θα οδηγήσει ενδεχομένω στην επιβολή κυρώσεων. Η Επιτροπή όμως θα κάνει μια σύσταση λέγοντας ότι ένα κράτος μέλος παρεκκλίνει. Μιλάω για την προληπτική πλευρά, την προληπτικό σκέλος του συμφώνου. Θα πρέπει λοιπόν από το Συμβούλιο, ναι πράγματι το διαπιστώνουμε αυτό, θα πρέπει το κράτος μέλος αυτό να λάβει αποτελεσματικά μέτρα. Στα αγγλογαλλικά λέμε effective action. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ελήφθησαν οι αποφάσεις ιδέουσες. Και αν το Συμβούλιο δύο φορές με δική πλειοψηφία αποφασίσει ότι πρέπει κάτι να γίνει, τότε μόνο οι υπουργοί, το Συμβούλιο Υπουργών μπορούν με την ειδική, αντίστροφη ειδική πλειοψηφία μπορούν να επιβάλλουν κυρώσεις. Ποτέ δηλαδή. Γιατί είναι πολύ μεγάλος ο χώρος και μπορούν να βρουν τη θέση τους εκεί κάθε είδους ίντριγγες ώστε να μην τεθεί ποτέ το πραγματικό ζήτημα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ εκφράζω την προσωπική γνώμη και επαναλαμβάνω ε, και ίσως και το Μπενελούξ, αφού το Λουξεμβούργο έχει την προεδρία του Μπενελούξ αυτή την ε, εποχή. Εκφράζω αυτήν την άποψη λοιπόν. Οι τρει διακυβερνήσει του Μπενελούξ θα επανεισαγάγουν στη συζήτηση αυτή την ιδέα. Δηλαδή να προβλεφθεί η, πλειο... η ψηφοφορία με αντίστροφη δική πλειοψηφία. Για να υπάρχει απαιτούμενη αξιοπιστία στις προτάσεις επιβολής κυρώσεων που μέχρι δεν υπάρχει. Μιλώ πάντοτε, επαναλαμβάνω, για το προληπτικό σκέλος. Και πρέπει να το πω πιο κατηγορηματικά σε σχέση με το διορθωτικό σκέλος. Κυρία Πρόεδρε, για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θέλω να σας πενθυμίσω, δεν το ξέρει κανείς, στις 11 Φεβρουαρίου 2010 στην βιβλιοθήκη Σολβέ είχα προτείνει εξώματος στην κυβέρνησή μου στις 3 και 50. Όλοι ήταν αντίθετοι, τώρα είναι όλοι υπέρ. Άρα εγώ ήμουν λοιπόν που πρότεινα αυτή την πολύ συνετή και σοφή ε, πρόταση. Ξέρετε τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνει. Όπως ε, προβλέπετε η ομάδα Φοντρομπάη μάλιστα έχει εργαστεί πάρα πολύ καλά και δύο πρόεδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Θέλουμε να μειωθούν οι μακροοικονομικές ανισορροπίες ως το δυνατόν περισσότερο, ώστε αν υπάρξει μια ασυμμετρική κρίση, ένα ασυμμετρικό σοκ στο μέλλον, να μπορούμε να ανθεσταθούμε καλύτερα ως ομάδα. Και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι νέες διαδικασίες σε περίπτωση μείωσης ε, του ελλείμματος. Υπάρχει μια ειδική διαδικασία που συνέλαβαν ο κύριος Φον Ρομπάι και η ομάδα του. Αυτά κυρία Πρόεδρε έχω να πω. Μου είχαν εδώ προετοιμάσει 48 σελίδες να σας διαβάσω. Όπως καταλαβαίνετε βέβαια έκανα μια μικρή περίληψη για να έχετε και εσείς το χρόνο να μου κάνετε τις ερωτήσεις σας. Και όπως πάντα θα απαντήσω σε κάποιες από αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Thank um, Σας ευχαριστούμε πολύ και για τα προηγούμενα σχόλια ότι ήδη έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη για τους συντονιστές ώστε στην κοινοβουλευτική μας επιτροπή ακολουθούμε την ίδια κατεύθυνση. Έχουμε 14 που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο και έχουμε λιγότερο από 50 λεπτά. Αυτό σημαίνει 3 λεπτά για ερώτηση και απάντηση εκάστοτε με το CatchDI και έχουμε φτάσει. Λόλινγκ, Σφεν Γκίγκολ, Σιλβι Κούλαρντ, Ούντο Μπούλμαν, Ζαν Πολ Γκάουζε, Τζόγκο Φέο, Βέρνα Λάγκεν, Σόφιεν Φελτ, Μίγουελ Πόρτας, Ρόντι Κρατσα, Βουλφ Κλίντς, Βίκυ Φόρντ και Κόριν Βόρτμαν Κούλ. Και εσεί, Τάισεν, θέλετε και εσεί να προσθεθείτε. Η, από πλευρά σα, 15η ε, παρέμβαση. Ένα λεπτό ερώτηση, δύο λεπτά η απάντηση. Και θα σας διακόψω αν ξεπεράσετε το χρόνο. Φιλίπ, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Αν κατάλαβα αυτά που είπατε, έχουμε ελπίδες ε, η ευρωπαϊκή εκπροσώπηση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να αναβαθμιστεί. Δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις. Τι πιστεύετε για τον κίνδυνο να υπάρχει ε, και το προκυκλικό, η προκυκλική ίσως επίπτωση κάποιας κρίσης. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Επίσης, κάτι που αναφέρατε, αλλά θα ήθελα λίγο να είστε πιο συγκεκριμένος. Η κίνδυνη της πολιτικής της ΦΕΝΤΗ πρόσφατη απόφαση συγκεκριμένα, το λεγόμενο quantitative easing, η δεύτερη αυτή φάση της έκδοση αυτών των ομολόγων. Τι κίνδυνου ενέχει αυτό. Απάντηση, θα απαντήσω στον Φιλίπ ότι ίσως να φαίνεται παράλογο να επιβάλλει κανείς κυρώσεις επιβάλλοντας πρόστιμα οικονομικά σε κράτη-μέλη τα οποία δεν έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν. Εγώ πάντα θεωρούσα ότι ποινικέ ε, κυρώσει είναι μέρος του πυρηνικού οπλοστασίου, θέλετε. Και πρέπει να περιμένουμε πριν φτάσουμε σε αυτό το στάδιο. περιμένουμε λοιπόν να γίνει διαδικασία μέσω αυτή τη αντίστροφης ειδική πλειοψηφία ε, θα μπορούσαν τα κράτη-μέλη να διορθώσουν ε, τα κακό κείμενα πολύ νωρίτερα. Ενώ τώρα μπορούμε απλά και ε, όσο θέλουμε να οικοτολογούμε και να αναβάλουμε συνεχώς και, και να αναβάλουν και τα κράτη-μέλη την εξυγένση των δημοσιονομικών. και δεν θα ήταν καλό σίγουρα να πάρει η Ευρωομάδα κάποιες αποφάσεις ε, οι οποίες να μην είναι οι σωστές. Οι αποφάσεις ε, τώρα της ΦΕΔ, τώρα για να απαντήσω σε όλα θα έπρεπε να μιλάω για πολλή ώρα, δεν θεωρώ ότι είναι σωστή πάντως η απόφαση της ΦΕΔ. Καταπολεμούμε το χρέος με χρέος. και αναγορευόμαθε σε αυστηρό κριτή της ε, κινέζικης οικονομικής νομισματικής πολιτικής, ενώ σίγουρα κάνουμε ακριβώς το ίδιο, με άλλο τρόπο. Ακολουθούμε ακριβώς την ίδια πολιτική. Εγώ βλέπω πληθωριστικούς κινδύνους. Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ένα επιπρόσθετο πρόβλημα ρευστότητα στη ΣΥΠΑ και δεν πιστεύω ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις θα επενδύσουν περισσότερα και ότι οι αμερικανοί καταναλωτές ε, θα καταναλώσουν περισσότερα μετά τις ε, ληφθήσεις αποφάσεις. Αντίθετα βλέπω τον κίνδυνο να υπάρξει στροφή προς ε, τις αναδυόμενες χώρες ο όγκος της ρευστότητας να μετακυλθεί σε ώρες αυτές αφού δεν μπορεί να απορροφηθεί εκεί. Λοιπόν, η απόφαση της Fed νομίζω ότι θα πρέπει να εμπλουτιστεί και καλό θα ήταν ίσως να έχουμε ε, και κάποιες επεξηγήσεις περισσότερες για να μην έχουμε καμιά ανησυχία. Η Άστριντ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κρίμα που πρέπει να περιμένουμε Θα ξαναρχίσουμε, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι κρίμα κύριε Πρόεδρε που θα πρέπει να περιμένουμε τα απομνημονεύματά σας που ίσως χρειαστεί και να περάσει κάποιος χρόνος για να καταλάβουμε ποιοι είναι οι βαθιοί λόγοι ε, της απουσίας του Προέδρου του Eurogroup από την ομάδα των 20, από το G20, αλλά τέλος πάντων στη συζήτηση που γυρίζει γύρω από το ευρώ και το σύμφωνο σταθερότητα, έχουμε την ιδέα τη χρεοκοπία ουσιαστικά ενό κράτου μέλους που είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσατε να μας ε, εξηγήσετε με απλά λόγια γιατί εμείς ως βουλευτές ε, είμαστε λίγο καχύποπτοι απέναντι σε πολύπλοκες ιδέες. Τι θα μπορούσε αυτό να, να σημαίνει συγκεκριμένα. Και δεύτερο, είναι ευκταίος κατά την άποψή σα ένα τέτοιο μηχανισμό. Διάβασα ότι ε, ο πρόεδρος της ΕΚΤ είναι ιδιαίτερα δύσπιστος ε, και δεύτερον γνωρίζετε φαντάζομαι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι ένα σημαντικός παράγοντας στην όλη διαδικασία του Συμφώνου Σταθερότητας. Θα πρέπει να δούμε και την κατανομή εξουσιών, όπως είπατε και εσείς, μεταξύ Κομισιών και Συμβουλίου. Στην όλη αυτή πρόταση που έχει διατυπωθεί εγκρίνεται αυτή την εξέλιξη που πιστώνουμε και εμείς, δηλαδή ότι η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποσκοπούσε σε κάποιο είδους ισορροπία μεταξύ των θεσμικών οργάνων, Άστριτ, δεν θα υπάρξει χρόνος για απάντηση. Λυπάμαι, λυπάμαι, λέει Άστριτ. Είχα και άλλες ερωτήσεις zo Θα μεταφράσω τα Λουξεμβουργιανά για τους μη Η κυρία Πρόεδρος μου δίνει δύο λεπτά για μια ερώτηση, ενώ η Άστριντ μου κάνει 7 ερωτήσεις σε σχόλια. Άρα 22 λεπτά θέλω για να απαντήσω. Τέλο πάντων, για να ξεκινήσω με το ουσιώδες. Πράγματι, τα απομνημονεύματά μου ε, θα αργήσουν. Θα... Είμαι Πρωθυπουργό όσο ε, στο Λουξεμβούργο ε, συνεχίζεται κανονικά η δημόσια ζωή, αλλιώ θα καταφύγω στη συγγραφή. Είμαι υπέρ της δημιουργίας ενός μόνιμου μηχανισμού επίλυσης κρίσεων Όχι ότι μας κατέλαβε εξαπίνηση η ελληνική κρίση, αλλά είδαμε ότι είμαστε σε μια κατάσταση που βλέπουμε ότι ο μηχανισμός δεν εφαρμόζεται και δεν έχει τα αποτελέσματα που θα έπρεπε. Άρα πρέπει να δημιουργηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός επίλυσης κρίσεων. Σε περίπτωση μάλιστα ε, που υπάρξει και χρεοκοπία, πτώχευση ενός κράτους και αυτό να μπορεί να ληφθεί υπόψη. ξέρουμε ότι αυτό που δεν περιμένουμε φτάνει και συμβαίνει τελικά. Ε, αυτό είναι ο γενικό κανόνα. Άρα πρέπει να υπάρχει αυτό ο μηχανισμό. Είπατε θέλετε απλέ ιδέε. Σα δώσω κι εγώ απλή απάντηση λοιπόν. Θα ήθελα να εξετάσουμε από πιο κοντά τα διάφορα στοιχεία αυτού του μηχανισμού επίλυσης κρίσεων. Ναι, θα πρέπει να μιλήσουμε και για τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ναι, θα πρέπει να εξετάσουμε εκ του σύνεγγυς τη συμμετοχή στο μηχανισμό και στα σενάρια πύλησης κρίσεων και του ιδιωτικού τομέα. Αλλά ο κύριος Τρισέ δεν είναι κατά του μόνιμου μηχανισμού. Όπως και αυτός έτσι και εγώ προειδοποιώ ότι ναι πράγματι πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ε, ίσως και δύο φορές προτού υπαγορεύσουμε ότι σε κάθε περίπτωση κρίση θα πρέπει να συμμετέχει ο ιδιωτικός τομέας. Εάν στο 100% των περιπτώσεων επίλυσης κρίσεων ε, το δουν κατά 80% δεν προβλέπει την ε, ανάληψη ευθύνης ιδιωτικού τομέα, αλλά μόνο στο 20% συμμετέχει ο ιδιωτικός τομέας. Εγώ πιστεύω ότι οι τράπεζες και οι διάφοροι φορείς ε, του ειδικού τομέα θα πρέπει και αυτοί να πληρώνουν για να αναλαμβάνουν τι ευθύνε του. Να πούμε όμω ότι η Ευρωζώνη είναι η μόνη νομισματική ζώνη όπου εξάντε και απριόρι ο ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να συμμετέχει, μου φαίνεται λίγο ότι χρειάζεται πιο εντελεχή μελέτη. ο κύριος Τρισέ είναι ανεξάρτητος, εγώ είμαι πολιτικός και μπορεί να είναι ανεξάρτητος ο κύριος Τρισέ. Όταν όμως ε, τα πει η Γερμανία ή πει κάτι η Γαλλία, ε, δεν ε, θεωρείται ανεξάρτητος ο κύριος Τρισέ. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να προσέχουμε, γιατί πρέπει να προσέχουμε τις σοβαρές προτάσεις που ακούγονται και τις σοβαρές ιδέες. Πρέπει λοιπόν να τίνουμε δίκονους, ε, τουλάχιστον προσεκτικό ε, σε αυτά που λέει ο κύριος Τρίσε. Τώρα για τη συναπόφαση, ναι, πρέπει να υπάρχει συναπόφαση και κάποια ευρωπαϊκά συμβούλια έχουν την τάση να το λησμονούν ενίοτε. Εντάξει, μία ερώτηση καθένας παρακαλώ. Διαφορετικά οι τελευταίοι δεν θα μπορέσουν να διατυπώσουν ερωτήσεις και δεν θα τα ανέχτα λοιπόν. Θα ε, υπάρξουν κυρώσεις. Εσείς λοιπόν παρακαλώ. Κύριε Γιούνκερ. Έχω μία ερώτηση και αυτό, αυτή είναι αν δω την προπαρασκευή των εργασιών για την οικονομική διακυβέρνηση και δω τα στοιχεία για την Ελλάδα 130% κρατικό χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ. Αυτή τη στιγμή κόστος του μηχανισμού σταθεροποίησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 8% ετήσια. Spreads 10% αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το επίπεδο χρέους θα απαιτούσε 10% του ΑΕΠ για να εξυπηρετηθεί. Πώς υπό αυτούς τους όρους μια χώρα μπορεί να διατηρήσει και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της. Δεν χρειαζόμαστε μόνο θεωρητικά αλλά και πολύ συγκεκριμένα χειροπιαστά για αυτές τις χώρες που βρίσκονται σε υπερβολική υπερχρέωση κοινέ διαρθρωτικές λύσεις <clears throat> που θα αντιμετωπίζουν το υπερχρέο ώστε να μπορέσουν να το αποσβέσουν. Θα με ενδιαφέρει η προσωπική σα άποψη πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Ευχαριστώ. Πολύ προσεκτικά λοιπόν και επισημαίνεται ότι θα πρέπει και εδώ προσωπικά να υπάρξει τοποθέτηση επ' αυτού για το ότι οι Έλληνες είναι υπερχρεωμένοι και κυρίως αυτό σε σχέση με την Ευρωζώνη η στάση της Ευρωζώνης και των άλλων Ευρωπαίων είναι κάτι το δεδομένο το οποίο συνοδήγησε σε αυτή την κατάσταση. Όμως αυτό δεν μπορεί να μας κάνει να απεμπολίσουμε αυτό το πρόβλημα το οποίο είναι πρόβλημα όλων μας. Η ελληνική κυβέρνηση που το θάρρος της θέλω να το υπογραμμίσω για άλλη μια φορά και να τονίσω ότι είναι θαραλέα και γενναία με τους όρους και προϋποθέσεις που από την Ευρωομάδα είχαν τεθεί είπε ότι ήταν σύμφωνη και πρέπει κανείς να υποθέτει ότι η άποψη της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι θα μπορέσουν να ανταποκριθούν ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν την κατάσταση και το χρέος. Και ξέρουμε ότι δεν είναι καθόλου απλό εγχείρημα αυτό. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει το θέμα του μηχανισμού κρίσης να το δούμε σε σχέση με την ερώτησή σας. Και πάλι με ιδιαίτερη ένταση Θέλω να πω ότι αυτά που είχα εγώ ε, προαναφέρει σε σχέση με τις ε, λύσεις από πλευράς ε, Ευρωζώνης, ουσιαστικά πιστεύω ότι αν και όταν θα έχουμε ένα μόνιμο τέτοιο μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσης ή αν θέλουμε να προσανατολιστούμε προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να ανασχοληθούμε με αυτά τα θέματα. Θα το κάνω εγώ αυτό, αλλά δεν έχω ακόμα εντολή της Ευρωομάδας για κάτι τέτοιο και είμαι κάπως επιφυλακτικός ώστε να προχωρήσει αυτό το θέμα ε, χωρίς, ε, οποιασδήποτε, ε, χωρίς οποιουσδήποτε όρους και σε σχέση και με τη χώρα μου. Με, πρέπει να δεχτούμε ότι υπάρχουν και όροι και κανόνες και περιορισμοί. Παρόλα αυτά είμαι πρόθυμος με τα ευρωομόλογα, είμαι ευγνώμων για το ότι προχωρεί αυτή η ιδέα και μια υποεπιτροπή θα πρέπει να συγκροτηθεί ώστε νυφάλια πέρα από κάθε δημοσιότητα και εντυπωσιασμό να ασχοληθεί με το θέμα των ευρωμολόγων και του τι μπορεί να γίνει. Αλλά με το Think Tank, με την ομάδα προβληματισμού θα πρέπει να προχωρήσει ώστε να δούμε πώς μπορούμε να χωρίσουμε τις, ε, το χρέος ε, των ε, χωρών σε, με κόκκινες ή γαλάζιες γραμμές και θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουν να βοηθηθούν αυτές οι χώρες και να μην εγκαταλειφθούν μόνες τους και να μην ε, απεμποληθούν αυτά διαβάζοντας σε σχέση με τα δημοσίευματα του τύπου ότι οι Γερμανοί λένε δεν είναι δυνατόν να είναι πάντα εκείνοι που θα πληρώνουν τα σπασμένα. Πρέπει να το πούμε λοιπόν αυτό σε σχέση με τους Λουξεμβούριους που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Αλλά πολλά πρέπει να μας προβληματίσουν. Ακόμα και η αφαίρεση του δικαίωματος ψήφου. Πρέπει να πω ότι δεν είναι δυνατόν να σκεφτόμαστε το αδύνατο. Πρέπει πρώτα να σκεφτούμε το εφικτό και το δυνατό και μετά το ανέφικτο ή το αδύνατο. Ευχαριστώ. σύμφωνο συνολικά ο μακροοικονομικός συντονισμός. Ελπίζω ότι δεν θα είναι κάτι το, κατά το μάλλον ή των αυτόματες κυρώσεις που θα υιοθετούνται, αλλά θα πρέπει με ευφυή τρόπο να δράσουμε benchmarking και πρέπει εδώ να διαπιστώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ναι μεν συνολικά έχει μια υγιή θέση εξωτερικού εμπορίου, αλλά υπάρχουν μεγάλες δυσαναλογίες και μη ισορροπές σχέσεις. Αν δει την ξεχωριστή θέση κράτους ε, και κράτους ξεχωριστά εκάστοτε μεμονωμένα. Τι γίνεται σε σχέση με τις ε, ε, τι ανισορροπίες αυτές. Ποια είναι η άποψή σας. Είναι ένα θέμα αυτό και ακούει κανείς διαφορετικές απόψεις και για τις μη ισόρροπες σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών. Μόνο τα ελλείμματα διαδραματίζουν ένα ρόλο ή και τα πλεονάσματα. Και πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μη ισόρροπη σχέση. Ποια θα ήταν μια λογική θέση και τι θα προτείνατε εσείς να γίνει για να είναι πιο υγιή τα πράγματα. Ευχαριστώ. Γενικά, Πρόεδρε, πιστεύω ότι παρότι υπάρχουν μη ισόρροπες σχέσεις και μέσα στην ίδια την Ευρωζώνη, δεν θα πρέπει σε αυτό το ληστηρό πεδίο να περάσουμε και να τραβηχτούμε σε αυτό από τους Αμερικανούς με τη δική τους δράση. Οι Αμερικανοί δεν έχουν μόνο ένα πρόβλημα ε, σε σχέση με την Γερμανία. Υπάρχει η Ευρωζώνη στις διατλαντικές σχέσεις και ο χώρος του δολαρίου. Και θα ήθελα να παρακαλέσω τους Αμερικανούς μας φίλους όταν πρόκειται για μη ισόρροπες σχέσεις και για την ισορροπία των πληρωμών, των, τους ισολογισμούς, να λάβουν υπόψη ότι σε σχέση με, αυτό το νόμισμα έχουμε από την 1η Ιανουαρίου 17 χώρες που συμμετέχουν σε αυτή την Ευρωζώνη και θα πρέπει στον Ευρωχώρο να, να δούμε ποια είναι η αναλογία και οι σχέσεις σε σχέση με το δολάριο Αμερικής και όχι να έχουμε κάποιες ξεχωριστές θέσεις που θα επηρεάζουν από πλευράς Αμερικανών τα πράγματα. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει εσωτερικά να το λάβουμε αυτό υπόψη. Σαφές αυτό λέει ο μιλητής και δεν έχω διαφορετική άποψη. Αλλά εσωτερικά δεν δημιουργούνται δυσκολίες για το ότι έχουμε διαφορετικούς απολογισμούς και ισολογισμούς. Τι θα πρέπει να γίνει. Ναι, το θεωρώ ότι μεσοπρόθεσμα είναι ένα πρόβλημα που δημιουργείται και στην Ευρωζώνη αλλά και σε σχέση με την ομάδα Φαν θα πρέπει πιο έντονα να ασχοληθούμε και με την ανταγωνιστικότητα και αυτό να δούμε ότι θα πρέπει να μας απασχολεί μόνιμα, αλλά δεν θα πρέπει να λέμε ότι ήρθε η συντέλεια του κόσμου. Θα πρέπει να σφιγμομετρήσουμε τα πράγματα μεταξύ μας, Αμερικανοί και Ευρωπαίοι, να δούμε τι θα γίνει σε σχέση με τις εξαγωγές και την τόνωση της οικονομίας μέσω των εξαγωγών, να υπάρξουν ισόρροπες σχέσεις και ισορροπίες που θα δημιουργηθούν και να υπάρξει τάξη πραγμάτων από πλευρά της Ομοσπονδιακής Γερμανίας και τόνωση της εσωτερικής ζήτησης. Να το τονίσω αυτό, ότι ενάντια στις προσδοκίες δεν είναι μόνο οι εξαγωγές αλλά και η εσωτερική ζήτηση που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από πλευρά τη ε, οικονομία τη Δυτική τη Ομοσπονδική Γερμανίας. Και αυτό εσωτερικά θα πρέπει να το διαβουλευτούμε εμείς. Δεν οφείλουμε ε, να λογοδοτούμε έναντι των ε, Αμερικανών λόγω των δυσαναλογιών που υφίστανται. τους εκτιμώ του Αμερικανού σίγουρα, αλλά τα πλεονάσματα δεν είναι δυνατόν ε, με κυρώσεις ε, να τιμωρηθούν. Και όποιος έχει πάνω από 4% πλεόνασμα σήμερα γίνεται ύποπτος αυτόματα και αυτό δεν θεωρώ ότι είναι εφικτό και δεν νομίζω ότι πρέπει να συνεχιστεί. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε τα αίτια αυτών των πλεονασμάτων και να δούμε σε σχέση με την θετική εκπροσώπηση αυτών των πλεονασμάτων να μην αντιμετωπίσουμε συμπτώματα μόνο και προσπαθήσουμε να θεραπεύσουμε συμπτώματα αλλά τα αίτια, να αντιμετωπίσουμε τα αίτια στη ρίζα τους ώστε αυτή η κατάσταση να μην διαιωνίζεται. Ευχαριστώ. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Président. Κύριε Πρόεδρε, Γιούνκερ, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση η οποία αφορά το κριτήριο του χρέους σε σχέση με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Τα κράτη γνωρίζουμε ότι πρέπει να διατηρούν εντός κάποιων ορίων το χρέος, αλλά πολλά το υπερβαίνουν αυτό το επίπεδο. Θεωρείτε ότι είναι ποσοτική η υποχρέωση. Όταν όμως ε, έχουμε μια περίοδο λιτότητας, θεωρείτε να αλλάξει αυτό το ε, ποσοστό γιατί κάποιες χώρες δυσκολεύονται. Ακούστε, για αυτή τη μείωση το 1.20, που να είναι μια κανονική διαδικασία για τα κράτη-μέλη δεν υφίσταται, είναι μια πρόταση ακόμα. Ούτε το Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο Υπουργών έχουν μέχρι τώρα καταλήξει σε συμφωνία. Άρα ε, δεν μπορούμε να αναλύσουμε λεπτομερέστερα την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρ' όλα αυτά μου φαίνεται ευστοχή και λογική. Πρέπει να υπάρξει σταθεροποίηση των δημοσιονομικών, σταθεροποίηση του προπολογισμού και τα κράτη που προσθέτουν χρέος στο χρέος ουσιαστικά αυξάνουν το δημόσιο χρέος τους, άρα θα πρέπει κατεπηγόντως ε, να προχωρήσουν στον τομέα της σταθεροποίησης 10-20 χρόνια σταθεροποίησης ε, στην Ευρώπη και αν θέλουμε να διατηρήσουμε τις, ε, τα δικαιώματα των επόμενων γενεών θα πρέπει να μειώσουμε τα επίπεδα χρέους. Παρατηρώ επίσης ότι αν το 2005 επί προεδρίας δεν είχαμε ε, κάνει κάποιες αλλαγέ στο σύμφωνο σταθερότητα πολλά κράτη της Ευρωζώνης θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να πληρώνουν πρόστιμα, να εφίστανται κυρώσει. Είχαμε μελετήσει τις οικονομικές συγκυρίες και δεν θέλαμε να επιβάλλουμε, να τιμωρούμε τα κράτη-μέλη μέσω του Συμφώνου σταθερότητα. αλλά αν δεν είχαμε κάνει τις ε, προτάσεις αυτές και τότε μάλιστα είχαν ε, ασκηθεί έντονες κριτικές. Τώρα, αν δεν είχε γίνει αυτό, πολλά κράτη, όπως είπα, θα πλήρωναν. Μία χώρα της ε, ζώνης του ευρώ δεν έχει υποβληθεί στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και αυτό αποδεικνύει ότι αν τελικά εφαρμόσουμε μια δημοσιονομική πολιτική σοβαρή τότε μπορούμε να το αποφύγουμε. Μιλάω για μια χώρα ε, που είναι ένα μικρό δουκάτο γύρω γύρω από κάποια μεγάλα κράτη. Ε, Herr Ευχαριστώ. Φυσικά και περιμένουμε ερμηνεία τα απομνημονεύματά σας, αλλά πριν από αυτό θα ήθελα να τονίσω το εξής. Η Σύνοδος Κορυφής του Ντοβίλ στη Ομάδα Εργασία του Ρομπόη υπήρχαν 20 ανοιχτά ερωτήματα για τα ζητήματα αυτά του ε, Ντοβίλ. Και τελικά δεν υπήρξε καμία ε, συμφωνία. Εσείς είπατε για να... Μίλησατε για κάποια αυτόματη επιβολή κυρώσεων. Υπάρχει μια σχετική πλειοψηφία ώστε οι αποφάσεις ε, της ομάδας Φόνο Ρομπάι να θεωρούνται έκφραση άποψης, όχι όμως μια οριστική λήψη απόφασης. Για πτώχευση τώρα, όταν μιλάμε για πτώχευση κάποιου κράτους. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο, ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Και θα πρέπει και οι πιστωτές να έχουν ε, λόγο. Αν δει κανείς τι έγινε στις Ηνωμένε Πολιτείες, μετά τις εκλογές πρέπει να δούμε πώς αποδίδει το νομοθετικό έργο. Θα πρέπει ίσως λοιπόν και οι πιστωτές ε, να συμμετέχουν κατά κάποιο τρόπο wir saßen in der van gruppe war ich auch als eurogruppen obermufti dabei an einem montag Ακούστε, εγώ ως επικεφαλής της Ευρωομάδας ε, ήμουν και εγώ ε, στην ομάδα Van Rompuy, στον Τοβίλ και προσπαθήσαμε να βρούμε λύσεις. Παραδείγματο χάρη, συμφωνήσαμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός επίλυσης κρίσεων Είπαμε επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει και αυτό να λαμβάνει απαραίτητα μέτρα για να μην παρεμβαίνουν κάποιοι εξωτερικοί παράγοντες. Επειδή ε, εσείς ε, μιλάτε για αυτούς που και είστε υπέρ του αυτοματισμού και ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σωστοί κτλ. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν οι αυτόματες αυτές κυρώσεις η ομάδα Φων έχει εκθέσει και τους λόγους γι' αυτό. αν όμως ε, παραμείνει ο μηχανισμός αυτός που μίλησα πριν αυτή η πλειοψηφία όσοι έχει, δεν πρόκειται ποτέ να καταλήξουμε σε επιβολή κυρώσεων. Ελπίζω να καταλήξουμε σε κάτι πιο λογικό. Σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητα, ε, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, αλλά σε ό,τι αφορά αλλαγή τη συνθήκη τώρα, αυτό θα πρέπει να γίνει κατά τρόπο που να μην δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Και δεν έχει να κάνει με την Βρετανία αυτό, αλλά με αυτούς που συναποτελούν την ομάδα του ευρώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πτώχευση, ενδεχόμενη πτώχευση κάποιου κράτους, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι δυνατόν να υπάρχει συμμετοχή των πιστωτών. Όχι φορολογούμενοι μόνο να είναι αυτοί οι οποίοι θα φέρουν το βάρος. Προσοχή όμως. Το να ξεκινήσουμε όμως από την ιδέα ότι θα υπάρχει 100% συμμετοχή σε κάθε περίπτωση, δηλαδή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, αυτό θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις ό,τι αφορά τις επενδύσεις και τους Ευρωπαίους επενδυτές. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να διευκρινιστούν οι αρχές και θα πρέπει να ακουστεί ο κύριος Τρισέ και όχι μόνο όταν μας αρέσουν αυτά που λέει. Um, uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιούνκερ και πρέπει να πω ότι μου άρεσαν πολύ αυτά που είπατε για τον αυτοματισμό και νομίζω ότι οι περισσότεροι που μίλησαν ε, είναι υπέρ αυτού, του, αυτής της αρχής αυτόματη επιβολή κυρώσεων δηλαδή. Θα ήθελα να μου πείτε τι πιστεύετε για το εξή θέμα. Στην Ευρώπη πολλές φορές ε, μας αποσπά η λεπτομέρεια και χάνουμε την ουσία. Το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να συμφωνήσουν για ε, τον αυτοματισμό αυτό οδηγεί όχι μόνο σε αυτό που είπατε εσείς, ότι τελικά ποτέ δεν θα επιβληθούν ε, κυρώσεις, όπως και το περιβόητο άρθρο 7 της Συνθήκης της Νίκαιας δηλαδή, αλλά δείχνει επίσης ε, κάτι πολύ επώδυνο, την έλλειψη πολιτικής βούλησης. Και αυτό θα έχει ένα πολύ αρνητικό ψυχολογικό αντίκτυπο και στο κοινωνόμισμα. Γιατί αυτό το βλέπουν όλοι. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη φαίνεται να μην μπορούν να αποφασίσουν ακόμη και όταν η κρίση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Ή δεν σας κατάλαβα ή δεν με καταλάβατε ή δεν κατάλαβα αυτό που δεν καταλάβατε. Τέλο πάντων, θέλω να πω, όταν μίλησα για τον αυτοματισμό τη επιβολή κυρώσεων, εγώ είπα ότι θα πρέπει στι κυρώσει αυτέ ε, ε, να συμπεριλαμβάνεται και η αφαίρεση του δικαιώματο ψήφου. Όχι, όχι, εγώ είπα ότι συμφωνώ για τις παρατηρήσεις, με τι παρατηρήσει σα για τον αυτονομισμό. Δεν μίλησα καν για δικαιώματα ψήφου. Είπα ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να αποφασίσουν για αυτόν τον αυτοματισμό και αυτό δείχνει έλλειψη πολιτική βούληση για ενίσχυση του συμφώνου. Αυτό είπα. Α, επειδή είπατε για το άρθρο 7, εμπερδεύτηκα, λέει ο κύριο Γιούνκερ. Και κάτι θεώρησε ότι κρύβεται πίσω από αυτά που ε, λέτε. Λοιπόν, ακούστε, ναι, αλλά νομίζω ότι έχουμε ε, πλειοψηφία, δηλαδή τα περισσότερα κρατημέλη θέλουν τα, τον, ε, τις αυτόματες κυρώσεις. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως. Για να εξευρεθεί συμβιβασμός, σε ό,τι αφορά αλλαγή της συνθήκης, Κάποιοι θεωρούν ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουν την επιθυμία του για αυτόματες κυρώσει. Και πρέπει να σκεφτείτε ότι μιλάμε για διαδικασία συναπόφασης. Δηλαδή, ακόμη και τα μέλη τη Task Force, τη ειδική αυτή ομάδα, εγώ ήμουν μέλο αυτή τη ομάδα, μπορούν, μπορούμε δηλαδή να επαναφέρουμε στη συζήτηση ένα σημείο από το οποίο το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εκφράσει την άποψή του και να συναποφασίσει, να δει πώς θα συναποφασίσει. Δηλαδή, απαρνούμεθα κάτι το οποίο θεωρούμε πρωτίστη σημασία επειδή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πήρε μια διαφορετική απόφαση. Ενώ γνωρίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται εδώ για να φέρει τον κοινό νου πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Νομίζω ότι πρέπει να επικαλεστούμε τον κοινό νου. Ναι, συμφωνούμε σε αυτό, λέει η Πρόεδρος. Μιγγέλ. Κύριε Γιούγκερ, Μιλήσαμε διαμακρών για τους αυτοματισμούς και τις κυρώσεις. Αυτό το οποίο διερωτώμε είναι το εξής. Αυτοματισμός σημαίνει ότι τα αίτια που προσδιορίζουν ένα πρόβλημα δεν λαμβάνονται υπόψη. Της προάλλης η κυρία Μέρκελ μιλούσε για την επίπτωση, για τη συμμετοχή των ε, πιστωτών για την επίλυση των ε, κρίσεων. Η πρώτη επίπτωση ήταν ότι αυξήθηκαν ε, τα επιτόκια στα ομόλογα της Πορτογαλίας. Δεν υπάρχουν κυρώσει για τι δηλώσει τη κυρία Μέρκελ ή για τι δηλώσει τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή ενό εκπροσώπου τη Κομισιόν. Διότι αλλιώ πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Υπάρχουν αυτοματισμοί για να αντιδρούμε κατά τη ανευθυνότητα, ναι ή όχι. Και τώρα έρχομαι σε ένα πρακτικό ερώτημα. Το πορτογαλικό χρέος το 2010 θα αγοράσει το σύνολο του χρέους αυτού με ένα δάνειο της τάξης του 1%. Ένας μηχανισμός που πραγματικά δεν καταλαβαίνω που έχει μια οικονομική λογική. επανέρχομαι στο θέμα της ελεγχόμενης χρεοκοπίας, γιατί είναι κάτι το οποίο ε, είναι καινούριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουμε εμπειρία, ενώ το, νομισμα... Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει και εμπειρία και μηχανισμό. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να συνδυαστεί μηχανισμός διάσωσης από τη μια πλευρά και χρεοκοπία από την άλλη. Σε, σε ποιο στάδιο της διαδικασίας θα μπορούσε να έρθει η χρεοκοπία. Και δεύτερον, αυτή η δυνατότητα δεν θα επηρεάσει, όποια και να είναι, επιμήκυνση ή το haircut κυρίως, δεν θα επηρεάσει τις αγορές, δεν θα ανεβάσει τα spreads. Και ε, τέλος ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή αναφέρεται πολύ στον ευρωπαϊκό τύπο ότι η διαδικασία αυτή ε, θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ε, ποια είναι η δική σας άποψη.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 μικρόφωνο. Ε, Λυπάμαι, εντάξει. Κύριε Πρόεδρε, η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα Fed έλαβε κατεύθυνση για δύο μέτρα να δώσει κονδύλια στην αγορά ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η αγορά. Ξέρουμε ότι η Αμερικανή βιομηχανία έχει δύο δις. Δεν είναι ε, έλλειψη χρημάτων λοιπόν. Είναι η έλλειψη προθυμίας, η έλλειψη βούλησης μια και δεν υπάρχει η ε, κερδοφορία. Πολλές φορές ε, αυτά τα κονδύλια βρίσκονται σε αναδυόμενες χώρες, γιατί εκεί η κερδοφορία είναι πολύ υψηλότερη. Οι δυσαναλογίες και οι μη ισόρροπες σχέσεις εντείνονται έτσι και δεν απαμβλύνονται. Ερώτησή μου, πώς εξηγείτε εσείς και πώς βλέπετε εσείς αυτή την κατάσταση. Δεύτερον, με την εισαγωγή ενός ευρωομολόγου, με την ε, συμμετοχή από πλευρά οικονομίας σε ένα τέτοιο μέσο, θα πρέπει να υπάρξουν κάποια κριτήρια. Δεν θα μπορεί αυτόματα όλοι να συμμετάσχουν αλλά μόνο όταν κάποιοι όροι και προποθέσει υλοποιούνται. Ευχαριστώ. Να απαντήσω κυρία Πρόεδρε για το πρώτο σημείο για να τοποθετηθώ. Ε, έφτασα με καθυστέρηση. Ευχαρίστω όμω να αναφερθώ, μια και πάντα είσαστε έγκαιρα εδώ. Όπως και εσείς πιστεύω και εγώ ότι αυτή η απόφαση της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας της Fed δεν είναι σκόπιμη και δεν είναι θα έλεγα ε, χρήσιμη και για τους λόγους που εσείς προαναφέρατε. Το πρόβλημα της Αμερικανικής οικονομίας ε, δεν είναι έλλειψη ρευστότητας. Το αντίθετο, το πρόβλημα δεν θα μπορέσει έτσι λοιπόν να λυθεί με τη δημιουργία ολόκληρων βουνών χρεών και δεν είναι αυτό ε, το, νόημα του εγχειρήματο. Και συμμερίζομαι τώρα σε σχέση με τις επικρίσεις που ο φίλος ε, Wolfgang Schäuble στις επικρίσεις που έχει ε, διατυπώσει έναντι των Αμερικανών δεν θα βοηθήσουν καθόλου αυτά τα μέτρα. Το αναφέρω αυτό δεν είναι ευφιές αυτό το μέτρο. Έχει τεράστια προβλήματα η αμερικανική οικονομία και με αυτό το πρόβλημα θα είναι ακόμα πιο επιβαρημένη η κατάσταση στην Αμερική με την ε, δανειακή πολιτική, με την πολιτική πιστώσεων. Τώρα, το να σχολιάζει κανείς με αρνητικό τρόπο αυτή την απόφαση πρέπει να μας κάνει να δούμε ότι θα δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα από όσα προβλήματα θα λυθούν μέσω αυτής της απόφασης από πλευράς Αμερικανών. Και πρέπει να το πούμε αυτό. Και πρέπει πραγματικά να διεξαχθεί μια ολόκληρη συζήτηση για να αποσαφινιστούν όλα αυτά και να διευκρινιστούν. Η δεύτερη ερώτησή σας αφορούσε το ευρωομόλογο και κάποια κριτήρια που πρέπει να συνάπτονται αμήν για το ευρωομόλογο. Και δεν ήθελα να ξεπεράσω κάποια όρια, γι' αυτό δεν αναφέρθηκα σε αυτό πιο πριν. Ουσιαστικά όσον αφορά τον μηχανισμό κρίσης, συμφωνώ με τις προτάσεις που ο Βόλφκαν Σόιμπλε διατύπωσε και έθεσε στο παιχνίδι. Αλλά θα πρέπει επίσης και για τα ευρωμόλογα να προβληματιστούμε και με τέτοιο τρόπο να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να αναπτυχθούν ώστε το χρέος των κρατών μελών να μπορέσει μέσα σε ένα κοινοτικό χώρο, σε ένα κοινό χώρο να επιληθεί και να αποσβεστεί αυτό το πρόβλημα και από κοινού να μπορέσουμε να δράσουμε προς όφελός τους και να δούμε σε σχέση με τα τραβηκτικά δικαιώματα από πλευράς των κρατών ε, εκείνοι που θα έχουν τις ευθύνες θα πρέπει να επιληφθούν, να υπομισθούν αυτές τις ευθύνες για να μπορέσουμε με σωστή στοχοθέτηση να πούμε ποιες υποχρεώσεις θα υπομίζονται κράτη τα οποία θα συμμετέχουν και αν όλα τα κράτη θα μπορούν να συμμετέχουν, να συμμετέχουν και υπό ποιου όρους και προϋποθέσεις. Θα πρέπει να γίνει αυτό όλοι να κερδίζουν και κανένας να μην χάνει από αυτό το εγχείρημα, κανένας να μην είναι χαμένος. Θα πρέπει λοιπόν το παιχνίδι έτσι να παιχτεί με αυτούς τους κανόνες και κανονισμούς. Θα έλεγα μπορούμε να το κάνουμε αυτό, ώστε η Γερμανία να μην έχει την εντύπωση που θα αποκομίζει ότι εκείνη θα είναι ο μόνος που θα πληρώνει και θα πληρώνει πάντα τα σπασμένα και εκείνοι θα πληρώνουν τις ζημιές των άλλων. Δεν πρέπει μια τέτοια εντύπωση να δημιουργηθεί εις βάρος των Γερμανών φορολογουμένων. Διαβάζω και ε, βλέπω ολόκληρο κύμα οργής και οργισμένων τοποθετήσεων που αρνούνται οι Γερμανοί να κάνουν κάτι τέτοιο. Δεν συμβαίνει όμως κάτι τέτοιο. Δεν θα είναι εκείνοι που θα πληρώνουν τα σπασμένα. Θα μπορούσα να τα έλεγα αυτά, αλλά δεν θα το κάνω. Right. Okay, we're now at the point. Λοιπόν, τώρα, εάν ε, είχαμε ξεκινήσει στις 3 και όχι στις 3 και 10, δεν θα είχαμε πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν θα κλέψω το δεκάλεπτο αυτό από την υπόλοιπη συνεδρίαση, ελπίζοντας να μείνει βέβαια και ο κύριος Γιούνκερ. Θα δώσω τώρα το λόγο στη Βίκη. Με λίγο διαφορετική ερώτηση, κύριε Γιούνκερ. Στην εισαγωγική σας ομιλία μιλήσατε για τη σημασία της διαχείρισης του υπερβολικού χρέους ε, και σε ό,τι αφορά το χρέος των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Και ακριβώς ε, γι' αυτό και η Βασιλεία κάνει νέε ε, συστάσεις για τις τράπεζες. Επίσης μιλήσατε για τους Financial Times και ότι πρέπει να του διαβάζουμε στου σημερινού, δύο μεγάλε τράπεζε ζητούν αλλαγή των κανόνων τη Βασιλεία. και πάλι Πόσο σημαντικό νομίζετε ότι είναι για την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, η εφαρμογή ε, της Βασιλείας με συνεκτικό τρόπο σε ολόκληρο τον πλανήτη και πώς εσείς εξετάζετε το ενδεχόμενο μεμονωμένες χώρες στην Ευρωζώνη μπορούν να έχουν την ευελιξία να αυξήσουν το κόστος δανεισμού και έτσι να ελέγξουν ε, την προμήθεια πίστης στα σύνορά τους εφόσον ξέρουμε ότι προέρχεται πολύ χρήμα από παγκόσμιες ε, πηγές. Um, Κύριε Πρόεδρε, για να απαντήσω σε ό,τι φορά την πρώτη ερώτηση, νομίζω ότι όλοι μας θα πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια ώστε η Βασιλεία Τρία να εφαρμοστεί παγκόσμια και επί ίσης όρης από όλους τους ε, εταίρους. 17 χρόνια χρειάστηκαν για να τεθεί σε ισχύ Βασιλεία 2 και 2 χρόνια μόνο για τη Βασιλεία 3. Θα ήθελα λοιπόν και οι, οι Αμερικανοί εταίροι και φίλοι μας να συμφωνήσουν και να εφαρμόσουν πιο πολύ την Βασιλεία 3 από ότι τη Βασιλεία 2. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και το βασικό σημείο συζήτησης που θα πρέπει να έχουμε όταν θα συζητήσουμε το ζήτημα με τις αρχές τον είπα Για το δεύτερο σημείο, δεν έχω αποκρισταλωμένη άποψη και μια ξεκάθαρη απάντηση να σας δώσω. Δεν μπορώ να σας απαντήσω αν δεν έχω την εξοδότηση να το κάνω. Έχετε γραπτή διαδικασία στο Κοινοβούλιο. Αν υποβληθεί ερώτηση εγγράφο, λέει η τότε ίσω να μπορέσετε να λάβετε και απάντηση. Φιλική επιστολή μου αρκεί, λέει ο κύριο Γιούνκερ. Και θα ζητήσω από του υπαλλήλου τη Κομισιόν να προετοιμάσουν και την απάντηση. Λοιπόν, θα διανύμουμε την απάντηση και την ερώτηση βέβαια. Κορίν. Ευχαριστώ. Αυτό το απόγευμα οι προσωπικές σας απόψεις είναι οι πιο ενδιαφέρουσες σε αυτή τη συνάντηση και πρέπει να πω ότι ως εισηγήτρια για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ε, καλωσορίζουμε τις απόψεις σας ότι χρειάζεται με ένας ε, αυτοματισμός δράσεων στην πρώτη φάση, start phase ε, των διαδικασιών. Ο κύριος πρόεδρος Ρόμπα είχε δύο εξηγήσει γιατί αυτό δεν ήταν εφικτό ή γιατί δεν ήθελε προς αυτή την κατεύθυνση να πορευτούμε. Ο πρώτος λόγος ότι δεν είναι δυνατό να υπάρχει μεγαλύτερος αυτοματισμός μέσα στην σημερινή συνθήκη της Λισαβόνας λέει. Και το δεύτερο επιχείρημα που ανέφερε ήταν ότι ενδιαφέρεται σε σχέση με την αποδοχή των μέτρων αυτών από τα κράτη-μέλη και για την δημοκρατική νομιμότητα είναι σημαντικό να υπάρχει απόφαση Συμβουλίου, διότι περισσότερος αυτοματισμός σημαίνει ότι περιορίζονται οι δυνατότητες ε, του Συμβουλίου να αλλάζει θέση ή να παίρνει κάποιες αποφάσεις. Πώς θα μπορούσατε να σχολιάσετε αυτές τις απόψεις και σε σχέση με τη δημοκρατική νομιμότητα ή δημοκρατική λογοδοσία, τι πιστεύετε, έχετε κάποιες απόψεις για κάποιες άλλες εναλλακτικές δράσεις. Ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για παράδειγμα, είχε προτείνει να είχαμε ένα συμβούλιο πραγματογνωμόνων Sachverständigungsrat υπό τη μορφή του, του γερμανικού συστήματος ένα συμβούλιο σοφών ώστε εκείνοι να έχουν την εποπτεία της λειτουργίας του συστήματος και το πώς χρησιμοποιεί αυτό το χώρο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να έχω τα σχόλιά σας γι' αυτό. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω, Πρόεδρε, ότι ο κύριος Φαν αν είχε πει κάτι τέτοιο θα ήταν αυτό ε, θα μπορούσε αυτό να είναι σωστό. Δεν νομίζω να το είπε και με αυτόν τον τρόπο. Διότι οι υπέρμαχοι των περισσότερων αυτοματοποιημένων κυρώσεων θα θέλαμε αυτές οι αυτόματες κυρώσεις να λειτουργούν μόνο όσον αφορούν και τις, ε, τη σύμφωνη γνώμη των ε, ίδιων των κρατών μελών. Θα ήθελα λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα των πιο αυτοματοποιημένων ε, κυρώσεων υπό το άρθρο 6 της συνθήκης που προβλέπει τις ε, διατάξεις αυτές για την Ευρωζώνη, για τον χώρο του ευρώ. Διότι με το άρθρο 6 μπορούν τα κράτη-μέλη της ζώνης ευρώ να προχωρήσουν πολύ περισσότερο από ότι τα υπόλοιπα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι έχουν σχέσεις πολύ στενότερες από ότι εκείνες ε, που βρίσκονται στο επίπεδο των 27 κρατών μελών και ελπίζουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε και περισσότερα αλλά οπωσδήποτε αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε σχέση με τις ε, αυτόματες, αυτοματοποιημένες ακυρώσεις σε σχέση με το άρθρο 6 που αφορά την Ευρωζώνη και το Ευρώ συγκεκριμένα. Δεν είμαι υπέρ των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας λέγοντας ότι πρέπει να είναι τέτοια, τόσο αυτοματοποιημένες αυτές οι κυρώσεις ώστε να μην έχει λέγει το Συμβούλιο των Υπουργών. Δεν συμφωνώ με κάτι τέτοιο. Αποκλειστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή αποκλει αποκλειστικά ένα άλλο σώμα να μπορεί να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις επικυρώσεων. Δεν είναι κάτι τέτοιο εφικτό. Οι κυβερνήσεις έχουν λέγει ναι, επ' αυτού και το Κοινοβούλιο όταν έρχεται η ώρα να λειτουργήσουν αυτά τα πράγματα από πλευρά διεργασιών και αυτό έχει λέγει, έχει λόγο να αρθρώσει. Αν αποφασίσουμε ότι όλες οι φάσεις της διαδικασίας θα διέπονται από την ενισχυμένη πλειοψηφία και τότε θα μπορεί το να υπάρχει η συμμετοχή των, του Συμβουλίου. Όχι μόνο δημοκρατικά νομιμοποιούμαστε σε σχέση με την κανονική ενισχυμένη πλειοψηφία, αλλά έχουμε επίσης και δημοκρατικούς κανόνες και δημοκρατική νομιμότητα όταν αποφασίζουμε με την αντεστραμμένη ενισχυμένη πλειοψηφία. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτή την αρχή σε σχέση με την Ευρωζώνη ως θέμα αρχής. Δεν λέω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δίκιο ή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει δίκιο ή, ή κάποιοι άλλοι μπορεί να έχουν δίκιο. Η Μαριάν παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία και εγώ να παρέμβω. Κύριε Πρόεδρε της Ευρωομάδας, έχω το συμπέρασμα του Ευρωσυμβουλίου για αυτό το θέμα που το διάβασα και όταν βλέπω την αφαίρεση δικαιώματος ψήφου ως κύρωση, όταν το διάβασα αυτό, αυτό που σκέφτηκα ήταν ότι αυτή η ιδέα μπορεί να ενταφιαστεί αμέσως, Διότι κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να το αρθρώσουμε και να το διατυπώσουμε. Για κάτι τέτοιο θα έπρεπε να αλλάξει η συνθήκη όσον αφορά το σύμφωνο, τη συμφωνία του μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων. Εσείς το βλέπετε έτσι ότι θα έπρεπε να αλλάξει η συνθήκη λόγω αυτού του μηχανισμού επίλυσης κρίσεων. Πιστεύετε ότι τα μέλη του Συμβουλίου θα συμφωνήσουν και θα περιοριστούν σε κάτι τέτοιο ή πιστεύετε ότι θα πρέπει να ξαναξεκινήσει μια συζήτηση αναθεώρησης των συνθήκων όπου όλα θα επανεξεταστούν. Μαριάν, πρέπει να σου πω ότι είναι πολύ επικίνδυνο να διαβάζει σε περισσότερε τη μια γλώσσα τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γιατί θα δείτε ότι τα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά διαφέρουν μεταξύ του, ιδίω όταν ε, περιγράφουν αυτό στο οποίο θα πρέπει να συνίσταται η οικονομική διακυβέρνηση, που ούτε καν το έχουμε πει. Απλά ο ίδιος όρος ε, με τρεις ε, διαφορετικούς όρους ε, ανάλογα με τη γλώσσα έχει καταγραφεί. Καλό λοιπόν είναι να επικεντρωθεί κανείς σε μία μόνο γλώσσα, αλλιώς θα περιέλθει σε σύγχυση προσπαθώντας να κάνει συγκριτική λογοτεχνική ανάλυση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ερώτημα της Μαριάν, οφείλω να πω ότι την ιδέα αυτή της αφαίρεσης δικαιώματος ψήφου την έχω καταπολεμήσει. Προβλέπει το άρθρο το συγκεκριμένο ότι όταν επαντηλημμένος παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, μπορεί να το αφαιρεθεί το δικαίωμα ψήφου. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε, δεν μπορούμε μάλλον να υποβαθμίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτό το επίπεδο όμως. Άλλο να μιλάμε για παραβίαση του Συμφώνου σταθερότητα. Δεν είναι το ίδιο με παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν θα πρέπει να τα συγχαίρουμε αυτά τα δύο. Πρότεινα και έγινε δεκτή η πρότασή μου ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που είχε εκφράσει την πρόθεσή του ο Χέρμαν Ροφόμπρο πάει να μελετήσει το θέμα αυτό, να μην μελετήσει το θέμα στο σύνολό του, αλλά να μελετήσει μόνο για θέματα σχετιζόμενα με το ευρώ. Να μην μελετήσει το θέμα λοιπόν εάν ε, για θέματα δικαιωμάτων εργασίας ε, ή οτιδήποτε ή αμυντικά θέματα κτλ. πρέπει να τεθεί θέμα ε, άρσης δικαιώματος ψήφο αλλά μόνο για τα οικονομικά ζητήματα. Ήθελα να περιορίσω το πεδίο στο οποίο θα, πάνω στο οποίο θα σκεφτεί ο κύριος Φον Ελπίζω να μην βρήκε τίποτα γιατί ακόμη και περιορισμένο το πεδίο σε πτυχές σχετικές με την ΟΝΕ, πάλι δεν θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα αυτή. Αυτό το οποίο μακράν θα πρότεινα θα ήταν να γίνουν πιο αυτόματες οι κυρώσεις και οι διαδικασίες σε κάθε φάση για την, για την λήψη αποφάσεων. Ας αφήσουμε την πυρηνική βόμβα για το τέλος και ας βάλουμε κάποιες νάρκες στην αρχή. Ας εκραγούν ε, ε, κάποιες μικρές νάρκες για να μην μπούμε σε ένα τεράστιο ναρκοπαίδιο. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι η τροποποίηση των συνθήκων θα πρέπει να είναι ελάχιστη και να δίνει στον μόνιμο μηχανισμό επίλυσης κρίσεων μια νομική βάση που θα ανταποκρίνεται σε όλες τις σταγματικές ανησυχίες και θα πληρεί τα σταγματικά κριτήρια. Εγώ θα πρότεινα να μην ε, τεχθεί καν θέμα αλλαγή τη συνθήκη, αλλά τα συνταγματικά δικαστήρια ε, τα μελετούν πολύ ενδελεχώς και έχουν δίκιο αυτά τα θέματα. Γι' αυτό λοιπόν ε, καλό είναι να μην δημιουργήσουμε νέα εμπόδια από τα συνταγματικά δικαστήρια μίας ή περισσότερων χωρών. δεν θα αφορά το άρθρο 125 αλλά το άρθρο 122. Να συμπληρωθεί δηλαδή το άρθρο αυτό με μια φράση που θα ανοίγει το δρόμο για τον μόνιμο μηχανισμό επίλυσης κρίσεων. Ή θα μπορούσε να μπει ε, κάτω από την ομπρέλα το 136 που αφορά την Ευρωζώνη. Κατά τα λοιπά θεωρώ ότι ο μόνιμος μηχανισμός επίλυσης κρίσεων θα πρέπει να περιορίζεται στην Ευρωζώνη και να μην επεκτείνεται συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας μην ξεκινήσουμε λοιπόν τη διαδικασία μιας ε, ανεφορίων ε, και περιορισμών ε, αναθεώρησης της συνθήκης. Σε αυτούς που δεν είναι υπέρ της συνθήκης της Λισαβόνας να μην τους δώσουμε δικαιώματα. Μικρή λοιπόν αλλαγή της συνθήκης, αλλά πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Αυτό θέλουμε.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 την ε, αναφορά που τον εισηγητή για την πρόοδο ε, και την ε, ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το IMF. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή η σειρά φτάνει στο τέλος της. Έχουμε την πρόταση οδηγίας για τη διαχείριση εναλλακτικών ταμείων. 30 Απριλίου 2009 σχετική ανακοίνωση και από τότε και μετά Πολλά έγιναν, έγινε πολλή δουλειά στο Κοινοβούλιο και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους, τους κοιόδης συγητές, οι οποίοι συνεργάστηκαν μαζί μου για το θέμα της διαχείρισης των κεφαλαίων εναλλακτικών επενδύσεων και εγκρίθηκε η έκθεση με πλειοψηφία. Βέβαια προσθέθηκαν και άλλα θέματα στη συνέχεια τα οποία θα πρέπει να τα διαπραγματευτούμε και να τα συζητήσουμε. Με τρεις προεδρίες συνεργαστήκαμε, την Τσέχικη, τη Σουηδική, την Ισπανική, αλλά και τη Βελγική Προεδρία. Η Βελγική Προεδρία μάλιστα πραγματικά με ιδιαίτερο ζήλο ασχολήθηκε για να προχωρήσει αυτό το θέμα σε επίπεδο των κρατών μελών, κάτι που δεν ήταν καθόλου εύκολο έγιναν έξι τριμερείς διάλογοι, ίσως και παραπάνω, όπου συμμετείχαν ε, οι διάφοροι πρόεδροι με τους συζητητές. Ανταλλάξαμε λοιπόν πληροφορίες και για την πρόοδο των εργασιών. Στις 17 Μαΐου του 2010 η, Επιτροπή μάλλον ε, πρότεινε, ψήφισε ένα σχέδιο έκθεσης. Ε, έγιναν μετά καμιά δωδεκαριά τριμερείς διάλογοι, πολύ εντυπωσιακό νούμερο εξίσου εντυπωσιακέ και 1690 τροπολογίε των συναδέλφων τη Επιτροπή. 12 περίπου λοιπόν τριμερεί διάλογοι, όπω είπα, ακολούθησαν. Έγιναν κάποιε καλέ και κάποιε λιγότερο καλέ συναντήσει, όπω είναι και το πεπρωμένο αυτών των δύσκολων διαπραγματεύσεων. Και στι 26 Οκτωβρίου, κατά τον τελευταίο τριμερή διάλογο, που το πρωί όταν ξεκινάγαμε δεν ξέραμε ότι θα είναι τελευταίο βέβαια, παρουσία του Didier Ρέντερ Υπουργού Οικονομικών του Βελγίου και Προέδρου του ΕΚΟΦΗΝ και του Επιτρόπου Μισελ Μπαρνιέ, καταλήξαμε σε συμφωνία για ένα συμβιβαστικό κείμενο, το οποίο θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια στις 11 Νοεμβρίου του 2010. 11 Νοεμβρίου είναι και η εκεχηρία Ίσως να μην είναι και κακή η χρονική αυτή σύμπτωση. Μετά λοιπόν από πάρα πολλές ε, τροπολογίες ε, ψηφίζουμε την ημέρα της ε, κεχηρίας. Καταφέραμε λοιπόν να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Λέω συμφωνία. Συμφωνία θα υπάρξει βέβαια μόνο αν την ψηφίσει το Κοινοβούλιο. Απλά στις 26 Οκτωβρίου καταλήξαμε σε ένα κείμενο που νομίζω ότι μπορεί να τεθεί σε ψηφοφορία χωρίς βέβαια να πω ότι όλα ε, είναι σύμφωνα με τις επιθυμίες μας. Θα ήθελα πάντως να ε, επιμείνω στο εξής. Τι πέτυχε το Κοινοβούλιο. Ίσως να μην φαίνεται άμεσα με την πρώτη ματιά. Στη Συμφωνία της 26 λέγεται ότι το κείμενο το συμβαστικό τροποποιήθηκε σε δύο-τρία σημεία, άρα δεν έγινε κάποια σημαντική τροποποίηση. Υπήρξαν, θα έλεγα, περιθωριακέ τροποποίησει εκείνη την μέρα, αλλά σημαντικέ γιατί είχαν να κάνουν με κάποιε διακήρυξει αρχή στι ιδεολογικέ σκέψει. Από την άλλη πλευρά, κάτι που μάλλον δεν έλαβαν υπόψη ορισμένοι εκτό του Κοινοβουλίου, είναι ότι υπήρξε προοδευτική πρόοδο μετά από του διαφόρου τριμερεί διαλόγου και χάρη στην αποφασιστικότητα των σκιωδών και του ηγητή ίσω είχαν αποτέλεσμα να υπάρξει, όπως είπα, πρόοδο σε κάποια σημεία. Θα τα αναφέρω. Πρώτα απ' όλα, το πολύ σημαντικό θέμα σχέσεις με τρίτες χώρες. Στην οδηγία έχουμε λοιπόν ένα διαβατήριο και σε ενδοευρωπαϊκό επίπεδο και από το 2015-2018 σε παγκόσμιο επίπεδο για τις τρίτες χώρες. Επίσης καταφέραμε να έχουμε μία εναρμόνιση των ελαχίστων ε, στις δημόσιες ιδιωτικές επενδύσεις ε, και έχουμε την αντικατάσταση κάποιων καθεστώτων από αυτό το διαβατήριο. Έχουμε επίσης αγάγει κάποιες διατάξεις οποίες δεν υπήρχαν στην αρχική πρόταση για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και δει ό,τι αφορά τους ε, κανόνες anti-stripping, μια επιχείρηση δηλαδή που εξαγοράζει μια άλλη να μην την κατακαιρματίσει, να μην την διαλύσει σε διάφορα κομματάκια. Άρα απαγορεύεται για δύο χρόνια να γίνουν κάποιες συγκεκριμένες ε, πράξεις. Επίσης, ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρείας στόχου είναι κάτι το οποίο πετύχαμε επίσης. Και κάτι άλλο που πετύχαμε στην τελευταία φάση των διαπραγματεύσεων ήταν μια ρήτρα αναθεώρησης για να μελετηθεί ο αντίκτυπος της οδηγίας σε περίπτωση στρέβλωσης ανταγωνισμού μεταξύ των Ευρωπαίων διαχειριστών και αυτών που έχουν την έδρα του εκτός Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε αφήσει κάποιο πεδίο σε ό,τι αφορά τις φορές διαχείριση παρά αυτά που επιθυμούσε το Κοινοβούλιο για κάποιου που θέλουν να έχουν την έδρα τους εκτός και η διαχείριση να γίνεται από φορεί οι οποίοι δεν αφορούνται από την οδηγία. Ασφάλεια επενδύσεων επίσης έχουμε σημαντικές ε, επιτυχίες και πληροφορίες ενημέρωση με περίπτωση μεταφοράς ευθύνης όταν έχουμε κατάσταση εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί έχουμε συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να υπάρχει ισοδυναμία. Σε ό,τι αφορά τους κανόνες οργάνωσης έγιναν συγκεκριμένε διευκρινήσεις. Για τη μόχλευση έχουμε κάποια κατόφλια με συγκεκριμένα κριτήρια για τους διαχειριστές και έλεγχος από τις αρχές. Επίσης παραπλεύρως επιτρέψαμε να υπάρξει πρόοδος με κάποια σχέδια της Κομισιόν ε, για, την πώληση, για τις ανοιχτές πωλήσει. και θα υπάρξει απαραίτητος ε, μηχανισμός ε, έλεγε η οδηγία, αυτό έχει πλέον αποσυρθεί γιατί ικανοποιήθηκαν τα αιτήματα του Κοινοβουλίου. Επίσης, ενίσχυση του ρόλου και των ε, αρμοδιοτήτων ε, του ΕΣΠΑ, κάτι το οποίο ήθελε το Κοινοβούλιο και νομίζω ότι και εκεί είχαμε πρόοδο. Επίσης, φροντίσαμε να ενισχυθούν οι εξουσίες του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στη διαδικασία έγκριση κατεξιοδότηση πράξεων από την Κομισιόν, ενίσχυση των υποχρεώσεων διαφάνεια απέναντι στι αρμόδιες αρχές και στου επενδυτέ ξεκίνησε και εδώ η προσπάθεια. Ό,τι αφορά τώρα την παθητική εμπορία, δεν καταφέραμε αυτό που θέλαμε στην αρχή. Δηλαδή, όχι τόσο την απαγόρευση αυτής, αυτού του είδους εμπορίας, κάτι που είναι δύσκολο να επιτευχθούμε, αλλά να υπάρχει αυστηρή πλαισίωση. Τουλάχιστον υπάρχει μια τολική σκέψη στην οδηγία, η οποία αναφέρει ξεκάθαρα ότι οι επενδυτές που επενδύουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ασκήσουν δέουσα επιμέλεια για να μην επενδύουν σε ταμεία που θα οδηγήσουν σε διευκόλυνση τη φόρο αποφυγής ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Επίσης υπάρχει μια διάταξη για τη ρύθμιση των επενδυτικών επιχείρησεων ε, που ε, διαθέτουν στο εμπόριο εναλλακτικά κεφάλαια, εναλλακτικέ επενδύσει. Υπάρχουν κάποιε μικρέ εξαιρέσει, υπάρχει όμω και η εισαγωγή τη αρχή τη αναλογικότητα ώστε η οδηγία αυτή που αρχικά κάπως αδιακρίτως ρύθμιζε οποιοδήποτε είδους ε, ταμεία που δεν ήταν ο PSVM, να προσαρμοστεί πλέον στο ε, στα διάφορα είδη πιστώσεων. Γιατί η κοινή βούληση του Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου ήταν κάθε οικονομική δραστηριότητα να ρυθμίζεται, να εποπτεύεται. Αυτό όμως συνεπάγεται ότι εφαρμόζεται η αναλογικότητα. Δεν μας ενδιαφέρουν δηλαδή πια μόνο οι συστημικοί κίνδυνοι, αλλά κάθε κίνδυνος που ενέχει μια οικονομική συναλλαγή. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους μας βοήθησαν στο έργο μας, φυσικά πάνω απ' όλα τους επιρογνώμονες ε, και το προσωπικό, του συνεργάτες της Γραμματείας Επιτροπής ΕΚΟΝ. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους γλωσσομαθείς υπαλλήλου και τους μεταφραστές. που πιέστηκαν λίγο από του εισηγητή γιατί έπρεπε να τηρηθούν κάποιες ε, προθεσμίες και ε, τους ε, υπόσχομαι να έχουν περισσότερο χρόνο για την επόμενη έκθεση. Uh,